ένα σημείο να συζητήσουμε για το Βόρειο Κάφκασο και κυρίως την περίπτωση του Όλεγ Ορλόφ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την παρέμβαση της κυρίας Χαουτάλα. Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα για την κατάσταση στο Βόρειο Κάφκασο και ιδίως για την περίπτωση του Όλεγ Ορλόφ είναι ε, ένα από τα πιο σημαντικά ψηφίσματα που, με τα οποία ασχοληθήκαμε στο Κοινοβούλιο. Η τραγωδία στο Βόρειο Κάφκασο έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, επηρεάζουν την καθημερινότητα στην Τσετσενία, στην ε, Ιγκετία, στη Βόρεια Οσετία. Οι παραβιάσεις δεν έχουν τελειώσει και μόνο πριν από λίγες εβδομάδες έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Κρόσνη, στο κοινοβούλιο της Τσετσενίας. 70 άτομα τραυματίστηκαν και οι περισσότεροι ήταν απλοί πολίτες. Στις 9 Σεπτεμβρίου 17 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο... στην ε, πρωτεύουσα της Βόρειας Οσετίας. Αυτές οι τραγωδίες του παρελθόντος ε, δεν έχουν ξεκαθαριστεί, κανένας δεν ξέρει ποιοι ένοχοι και τα θύματα δεν γνωρίζουν τι έγιναν στους αγαπημένους τους και στα παιδιά τους, πού πέθαναν, πού είναι τα σώματά τους και τα πτώματά τους. Ο φαύλος κύκλος της βίας και της ατιμορρησίας ε, έχει παραλύσει τη χώρα, αλλά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη βία οδήγησε σε ε, επιτάχυνση της ε, επιδείνωσης κατάστασης. Υπάρχει βέβαια το φάσμα του, της τρομοκρατίας και άνθρωποι εξαφανίζονται ακόμα και στην πρωτεύουσα, ε, ακόμα και στη Μόσχα δηλαδή, ακόμα και στην Αγία Πετρούπολη. και αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ε, η, ο, ο κύριος Ορλόφ κέρδισε το βραφείο Σαχάροφ το 2009 και αντιμετωπίζει ποινικές, ποινική δίωξη. Νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να πει φτάνει πια θα πρέπει μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης να ασχοληθούμε ε, για τα ένδικα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκοσο και για το πώς θα σταματήσουν αυτές. Κυρία Σάκη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα ο πρόεδρος Μπούζεκ ανακοίνωσε ποιο έλαβε το βιβλίο Ζαχάροφ για φέτος, το οποίο εκφράζει βεβαίως την ε, ελευθερία σκέψης και των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλώντας για το βραβείο Νόμπελ, ζήτησε από την Κίνα να απευθερθεί ο Λίντζιαμπο και είπε πως η ελευθερία δεν είναι απειλή, αλλά οι απειλές για την ελευθερία είναι πολλές. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που υπερασπίζουν ανθρώπινα δικαιώματα στο Βόρειο Κάυκασο. Το περσι... Ο Λεγκορλόφ, Σεργέη Κόβαλεφ και η Λουτμίλα Αλεξέγεβα που έλαβαν πέρσι το βραβείο Ζαχάροφ δεν μπόρεσαν να το λάβουν προσωπικά καθώς απειλεί τη ελευθερία τους. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σχέσεις με τη Ρωσία και εμείς και ο ΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε η Ρωσία έχει δεσμευτεί να υπερασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αλλά απέχουμε ακόμα πολύ από εκεί. Εκφοβισμοί, εξαφανίσεις, συστηματικές συμβαίνουν και δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης ούτε στο ίντερνετ. Έχουμε 20.000 περιπτώσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει πω δεν θα υπάρχει και σταθερότητα χωρί κράτο δικαίου. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τη Ρωσία να μην συμμορφώνεται με τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Αναμένουμε και θα φροντίσουμε οι εκπρόσωποι του Memorial να έρθουν σε αυτό το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο θα συμβολίζει την ελευθερία και τα δικαιώματα όλων των πολιτών του Νοτιοβόρειου ε, Βορείου Καυκάσου. Με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο είναι ο επόμενος μας ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ανησυχεί ιδιαίτερος ε, το κλίμα εκφοβισμού που επικρατεί στη Ρωσία εις βάρος των ακτιβιστών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας προς τον Όλε Κορλόφ, τον περσινό βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι από τις λίγες φωνές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συνεχίζονται οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δυστυχώς ε, οι άνθρωποι αυτοί ζουν με το φόβο καθημερινά. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους τρομοκρατία και ριζοσπαστικοποίηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί το κράτος δικαίου και τα μέσα που της προσφέρει το δίκαιο. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η καταπίεση και η καταστολή στο, στο Βόρειο Κάφκασο, αλλά να γίνονται πιο πολύ σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αν θέλετε δικαιοσύνη, θα πρέπει να έχουμε και υποκειμενική και ενδικειμενική διάσταση. Στο Βόρειο Κάφκασο αυτό σημαίνει θα πρέπει να, ότι θα πρέπει να παταχθεί η ατιμορρησία. Θα πρέπει οι πέτοι να παραπέμπονται στα δικαστήρια, να δικάζονται και να καταδικάζονται εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους. Επίσης θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των θυμάτων. Και να υποστηρίξουμε τον Όλεκ Ορλόφ αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και στις συνομιλίες μας με τη Ρωσία όταν συνάπτουμε σχέσεις με τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να επισημάνουμε στη Ρωσία ότι οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα αν θέλει να είναι πραγματικός εταίρος της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρ των δικαιωμάτων των λαών. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι ξεπέρασα το χρόνο μου, μίλησα 1,5 λεπτό. Ο κύριος Τσαρνέτσκι. Την εποχή του κομμουνισμού, όταν η Σολιντάρνο στην Πολωνία έδινε μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ακουγόταν το σύνθημα «Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς αλληλεγγύη». Στο σημερινό πλαίσιο ε, και με αυτά που συμβαίνουν στο, στη Βόρειο Κάφκασο αλλά και σε πολλές περιοχές της Ρωσίας θα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σταθερό ποιήση, δεν υπάρχει σταθερότητα χωρίς κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε αυτά υπόψη ταυτόχρονα. Γιατί κυρίες και κύριοι δεν μπορούμε τις ε, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μας με τη Ρωσία να τις ε, αντιμετωπίζουμε ως κάτι τελείως ξεχωριστό από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αλληλένδετες αυτές οι σχέσεις. Δεν πρόκειται για τελείως διαχωρισμένα ζητήματα. Είναι συγκοινωνούν δοχεία το οικονομικό, το πολιτικό σκέλος με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να, να εξασφαλίσουμε σεβασμό δικαιωμάτων, δικαιώματα ελευθερία έκφραση, για, πράγμα, για παράδειγμα. Θα πρέπει να απαιτήσουμε και από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχάροφ. Ένα πολύ σημαντικό βραβείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσαρνέτσκι. Η κυρία Βεριζιά, για 1,5 λεπτό. Merci, Monsieur le Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να κάνω μία ερώτηση προσθεί το βραβείο Ζαχάροφ, γιατί η κυρία Χάουταλα μα εξέφρασε τι ανησυχίε τη για την κατάσταση του κυρίου Ορλόφ. Ο κύριο Ορλόφ είναι από του τρει επικεφαλεί του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζαχάροφ, που βραβεύθηκε πέρυσι του κέντρου Memorial που βραβεύθηκε πέρυσι με το βραβείο Ζαχάροφ. Ήταν από τους ανθρώπους που τολμούν να στυλιτεύσουν την κατάσταση και να επισημάνουν την παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Πέρυσι είχαμε τη δολοφονία της κυρίας ε, Στεμίροβα που καταδίκασε και ο κύριος ε, Ορλόφ. Ε, δυστυχώς θεωρήθηκε αυτό συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Προέδρου Καντήροφ και ασκήθηκε μήνυση εναντίον του. Και μάλιστα πέρυσι ο κύριος Ορλόφ καταδικάστηκε και εμείς δεν είπαμε τίποτα. Στις 6 Ιουλίου κατηγορήθηκε και πάλι ο κύριος Ορλόφ και σήμερα απειλείται με τριετή ποινή φυλάκισης. Το βραβείο Ζαχάροφ θέλει να αναδείξει τον αγώνα των ανδρών και γυναικών που δίνουν μάχη για τη δημοκρατία και δίνοντα αυτό το βραβείο του έτουμε υπό την προστασία μα. Τι κάναμε όμω για τον κύριο Ορλόφ, τι κάναμε για αυτού που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και την Τσετσενία, πώ θα προωθήσουμε τον ε, διάλογο με την Ρωσία ώστε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βόρειο Κάφκασο. Θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε σιωπηλοί ένα χρόνο μετά την δολοφονία της κυρίας Στεμίροβα να μην ξεκινήσουν οι ποινικέ έρευνες. Ναι. Να εκφοβίζονται ή να εξαφανίζονται αντιφρονούντες ή ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς καμία νομική συνέχεια προς τι το βραβείο Ζαχάροφ, τι εξυπηρετούμε κι εμείς αν ανεχόμαστε τέτοιες παραβιάσεις δικαιωμάτων χωρίς να εμποδίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει αυτό το θέμα επιτάπητος, γιατί Καλό είναι να υπάρχει πρόοδο, αλλά όχι μόνο σε θέματα πέραν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει να υπαγάγουμε την δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα οικονομικά συμφέροντα ή τα πολιτικά συμφέροντα ορισμένων χωρών μελών, για να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να επιμείνουμε και είναι κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι στην αίθουσα σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσελτ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Βόρειος Κάφκασος ήταν θύμα τσαρικής απεικιοκρατικής πολιτικής και στη συνέχεια ακολούθησε και το σταλινιστικό καθεστώς αλλά δυστυχώς ε, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ε, υπήρξαν δύο ομοί και βίαιοι πόλεμοι σχεδόν ε, γενοκτονία των Τσετσένων και σήμερα μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια περιοχή ε, όπου ε, δορυφόροι της Ρωσίας τύπου Καντήροφ παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς καταδικάζουμε αυτά τα καθεστώτα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γι' αυτό, για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση, χρειαζόμαστε τα εξή τρία στενή συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς και οι διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται εκεί και προσπαθούν να αποκρούσουν ε, τη Ρωσία. Και εδώ έχει σημασία κομβική το memorial. Γι' αυτό ζητούμε για τον κύριο Λέγκορλοφ όχι να τον αφήσουμε αμέσω ήσυχο, αλλά και να τον υποστηρίξουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι πολύ αξιόλογη και αξιέπαινη η προσπάθειά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είμαστε στο πλευρό των λαών του Βορείου Καυκάσου και το οφείλουμε και στη συναγωνίστριά μας και φίλη μας Εσδεμίροβα που την ξέραμε πολύ προσωπικά και πλέον θα πρέπει η δολοφονία της να διαλευκανθεί. Το οφείλουμε αυτό στο Βόρειο Κάφκασο για να φροντίσουμε επιτέλους να υπερισχύσει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Λέγκορ Λόφ έχει δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Βορείου Καφικάσου είναι ότι οι πολιτικοί έχουν αγνοήσει το σημαντικότερο, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο έτσι μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Βόρειο Κάφκασο. Αλλιώς θα συνεχίσουν να στηρίζουν οι κάτοικοι την τρομοκρατία. Οι οργανώσεις όπως το Μεμοριάλ χρειάζονται υποστήριξη διότι ε, είναι απαραίτητες για μια σταθερή και δίκαια κοινωνία. Χρειάζονται λοιπόν την υποστήριξή μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επικρίνουμε οποιασδήποτε αρνητικές εξελίξεις και να εκφραστούμε υπέρ των θυμάτων απαγωγής ας ο κύριος Μύρισκη. Κύριε Πρόεδρε, στο ψήφισμα λέει ότι είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βόρειο Κάυκασο. Την περιοχή αυτή την ξέρω καλά. Δεν έχω πάει μόνο μία φορά, έχω πάει πανελειμμένα. Θα ήθελα να πω ότι οι αρχές της Τσετσενίας δεν έχουν κανένα δικαίωμα να καταδικάζουν τον κύριο Ορλόφ. Αν θεωρεί ε, η Τσετσενία ε, Μάλλον ο κύριος Ορλόφ θα πρέπει να αποδείξει τα δικαιώματά του και το δίκαιο του στο δικαστήριο, αν όχι στα ε, ρωσικά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς δεν θα πρέπει να έρθουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δικαιολογούμε μία πλευρά και να ε, ε, παίρνουμε θέση. Κάθε πλευρά θα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Και θα ήθελα να φροντίσει ο κύριος Ορλόφ να σκέφτεται πριν μιλήσει, γιατί και η συκοφαντία είναι αξιόπινη πράξη. Πρόκειται για ένα παράδοξο. Την ε, μέρα που αποφασίζουμε για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ το 2010 να μιλάμε για αυτήν ε, την ε, δίκη του κυρίου Ορλόφ που πήρε το βραβείο πέρυσι. Βραβεύθηκε πέρυσι ο κύριος Ορλόφ γιατί με τρόπο γενναίο πάλεψε για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των άλλων και στη Τσετσενία. Σήμερα ο κύριος ε, Ορλόφ διώκεται διώκεται για την ε, θέση του για την Τσετσενία. Η δίωξή του όμως ε, δεν θα υφίστατο αν από πίσω δεν υπήρχε η υποστήριξη της Ρωσίας. Πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση στον κύριο Μευδέιεφ για να σταματήσει η κατάσταση στην Τσεσενία. Η κυρία Μπασέσκου. Οι δημοκρατίες του Βορείου Καυκάσου είναι θέατρο βιαίων βιοπραγιών κάθε μέρα. Οι επιθέσεις κατά του, της Βουλής της δείχνουν ότι υπάρχει εκεί μεγάλη αστάθεια. 15 χρόνια μετά την έκρηξη των τσετσενικών πολέμων υπάρχουν ακόμη 8.000 εκτοπισμένοι και η τύχη των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας ανησυχεί υπάρχουν ε, καταδίκες αυθαίρετες και η περίπτωση του Ολέγκ Ορλόφ είναι μία από τις περιπτώσεις Ρώσων που δικάστηκαν για χωρίς ε, αποδείξεις όπως είχε γίνει και με την Εστεμίροβα το 2009. Οι έρευνες από το θάνατό της μέχρι τώρα για να διαβλευκανθεί αυτός δεν έχουν καταλήξει ακόμη πουθενά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι παραπάνω ώστε να διασφαλίσουμε δίκαιες έρευνες και για τα μέλη του Μεμοριάλ. Μάλιστα η κυρία Κορχόλα. Κύριε Πρόεδρε, ο Βόρειος ε, Κάφκασος ε, είναι γνωστός ε, για τις κρίσεις του. Έχει ο πόλεμος από την Τσετσενία, έχει επεκταθεί και στην Ιγκουσετία και στον Δαγεστάν. Εγώ δεν θα ξεκινήσω πολεμική για το αν είναι απολευθερωτικός αγώνας ή όχι. Η κατάσταση όμως είναι απελπιστική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς πέρυσι ε, δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ στην οργάνωση Memorial, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο Βόρειο Κάφκασο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κύριος Ορλόφ είναι αυτός που πήρε το βραβείο. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τα λόγια του. Εμείς γνωρίσαμε αυτόν τον κύριο ως προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο κύριος Λιβινέγκο που δολοφονήθηκε στην Αγγλία και η κυρία Στεμίροβα που επίσης δολοφονήθηκε, όλοι κατακρίθηκαν από την Ρωσία και μπορούμε εμείς να, έχουμε εδώ, να συντάξουμε έναν μακρύ κατάλογο των μη διερευνημένων δολοφονιών. Ο κύριος Σόνικ. Θα ήθελα Να αναφερθώ στην συνάδελφο η οποία είπε ότι δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ οι εκπρόσωποι του Μεμοριάλ για να πάρουν το βραβείο. Ε, δεν είναι δυνατόν. Πέρυσι ήρθανε και πήραν και το βραβείο. Η έκθεση που ετοίμασε η συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφερόταν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη ζώνη του Καυκάσου. Οι Ρώσοι όμως είναι αυτοί που παρεμποδίζουν στην ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άμαχοι απειλούνται. Βία, βασανιστήρια, κακομεταχείριση, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αυθαιρεσίες, αυθαίρετες συλλήψεις. Και οι οργανώσεις που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ε, έχουν καμία αποτελεσματικότητα στην περιοχή. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο Βόρειο Κάφκασο και να υπάρξει δημοκρατισμός ούτως ώστε να μην υπάρχει ατιμορρησία στην περιοχή. Η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΕ. Βλέπω τον κύριο Μικολάσικ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Βόρεια Κάφκασο είναι η αμέλεια και η αδράνεια του έξω κόσμου σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές όμως αποσταθεροποιούν την περιοχή και μειώνουν τις πιθανότητες βελτίωσης. Και ενθαρρύνουν και τον κύριο Καντήροφ, ο οποίος δεν σέβεται τίποτα ούτε νόμο, ούτε κανόνες, ούτε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, είναι δύσκολο να ενημερώνεται για όλα αυτά η κοινή γνώμη και δεν υπάρχει καν διαδικασία διαβούλευση συνεννόησης με την κοινή γνώμη. Αυτό ήθελα να αλλάξουν τα μέλη της οργάνωσης Memorial και από ό,τι φαίνεται ε, δυσκολεύονται πάρα πολύ και δεν ε, μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα πρέπει να ενημερωθούν για τα εκεί τεκτενόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέτσου. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου και ε, ε, όλη μας ε, την αγάπη να στείλουμε στην οργάνωση Memorial που μάλιστα πέρυσι κέρδισε το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Τσετσένος πρόεδρος και η νέα προσφυγή του στη δικαιοσύνη συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις και διώξεις των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το πιο κατάφορο γεγονός ήταν η δολοφονία της Νατάλια Στεμίροβα που ήταν επικεφαλής της Τσετσενικής Memorial. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ κατά της ατιμορρησίας των αυτοργών όλων αυτών των δεχτών εγκλημάτων γιατί θα πρέπει όλα αυτά να τα θέσουμε και υπόψη των ρωσικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ ταυτόχρονα παραλείπουμε τελείως το μεγαλύτερο από αυτά στον Βόρειο Κάφικαστο. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί οι Μοχαμπίτ που προέρχονται από έξω εκπαιδευμένοι και με πολύ συγκεκριμένους στόχους, με με συγχωρείτε, οι Βαχαμπίτες είναι άνθρωποι που χρηματοδοτούνται από τις ίδιες πηγές με άλλους τρομοκράτες. Και δυστυχώς στο ψήφισμα αυτό το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρεται με την παράληψη αυτής της διάστασης. Για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες συνθήκες. Αν υπάρχει χρηματική υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και υπάρχει, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε πια τίποτα. Και αυτό δεν το λέει το ψήφισμα. Υποστήριξα απολύτω ε, το ψήφισμα αυτό που υποστηρίζει και η πολιτική μου ομάδα και ζητεί ε, δράση για να υποστηρίξουμε τον Ολέγ Ορλόφ που έχει βραβευτεί με το βραβείο Ζαχάροφ και τι αξίε που πρεσβεύει και υπηρετεί στο Βόρειο Κάφκασο. Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό ότι καθόλου δεν θεωρώ την ομάδα μου ε, ότι ε, αντικατοπτρίζεται η θέση της στα λόγια του κυρίου Μίρσκι που ε, κατέκρινε τον κύριο Ορλόφ και είπε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιότητα που έχει το αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να καταφέρεται κατά του κυρίου Καντήροφ. Μα δεν χρειάζεται κανείς να είναι αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ανήκει στο Μερμόριο ή να έχει το βραβείο Ζαχάροφ για να έχει το δικαίωμα να επικρίνει οποιοδήποτε αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης. Κάθε χέφρον άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Ραούλ Ρωμέβα προηγουμένως και κάλεσε όχι μόνο το Κοινοβούλιο αλλά και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δουν την επικίνδυνη κατάσταση που αναπτύσσεται τώρα στη Δυτική Σαχάρα και να ζητήσει να παρεύουμε έτσι ώστε οι μαροκινές αρχές να μην ε, συλλαμβάνουν τους ή που ε, αγωνίζονται κατά της παράνομης κατοχής. Ο πρόεδρος διακόπτει συγγνώμη, αλλά μιλάμε για το Βόρειο Κάφκασο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επίτροπος, η κυρία Κόκκιγαν Κουίν. Uh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο. Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Τσετσενία θεωρήθηκε ότι έληξαν πέρυσι, αλλά οι βίες, οι βίες πράξεις συνεχίζονται και στην Ιγκουσετσία επίσης. Η ένοπλη επίθεση της Τρίτης κατά του, της Βουλής του Γκρόσνη μας θύμισε ότι η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και ασταθής. Η Αντιπρόεδρος Άστον, η εκπρόσωπος για τα εξωτερικά, έχει δηλώσει ότι Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την τρομοκρατική βία και τις επιθέσεις αυτοκτονίας. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων που ήταν απλοί πολίτες και δύο αστυνομικοί κατά την εκτέλεση του καθήκοντός των. Συνεχώς σημειώνονται βέβαια επιθέσεις και κατά των αγωνιστών των ανθρωπι... υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμεί αποτείωμε φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή του και συνεχίζουν την ε, δουλειά του υπέρ στον αγώνα αυτών υπό τέτοιε συνθήκε ανεξάρτητους δημοσιογράφους σε ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία που αντιμετωπίζουν πιέσει και βιαιότητε. Ο Λέγκορ Λόφ, επικεφαλή του Τμήματο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεμοριάλ και η κυρία Λουιτμίλα Αλέξη, Αδιλέξια, έχουν υποστεί τέτοιες πιέσεις. Ο πρόεδρος Καντήροφ κατηγορήθηκε, ε, κατηγόρησε τον κύριο Ορλόφ αλλά δεν έγινε τίποτα δικαστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την δεύτερη δίκη του κυρίου Ορλόφ. Το ίδιο κάνουν και άλλες οργανώσεις. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ μίλησε κατά του νομικού μηδενισμού που υπάρχει, που επικρατεί στη Ρωσία. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα σε συνεργασία και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ένωση θεωρεί πολύ σημαντική την ευκαιρία που έχει να συζητήσει αυτά τα προβλήματα με τις ρωσικές αρχές και Χαιρόμαστε για την ανοιχτή στάση που τήρησε ο πρόεδρος Μετβέντεφ ως προς τις σχέσεις του με την Ένωση για το θέμα αυτό. Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων συνοργανώνονται επαφές για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Η συζήτηση για τον Βόρειο Κάυκασο έχει λήξει. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε πρώτον έξι ψηφίσματα για τις βίες διώξεις στο Ζιμπάμπου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, πόχες, κρίνονται.